Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη τη συνεδρίαση ε, τη Επιτροπή Απολογισμού που είναι εξαιρετικά σημαντική σήμερα. Όλοι. Ξέρουμε ότι είναι ουσιώδου σημασία αυτό που θα συζητήσουμε. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Έτιγκερ που είναι εδώ με του συνεργάτε του. Του ευχαριστούμε για την αφοσίωσή του και τη δουλειά που έχουν κάνει ω τώρα η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προπολογισμό δεν οδήγησε σε αποτέλεσμα. Μείναμε σε αποτυχία. διότι το Συμβούλιο προέβλεψε ένα δις για την Τουρκία και την υποδοχή των προσφύγων εκεί, ε, σύρων προσφύγων. Και θεωρήσαμε ότι αυτή είναι μια χειρονομία αρνητική ως προς το Κοινοβούλιο που δεν είχε δικαίωμα έκφρασης. Ζητήσαμε λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες και οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναζήτηση εξισορρόπησης της όλης κατάστασης εκτίμησε ότι είναι στιγμή να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 15.3 του Δημοσιονομικού Κανονισμού. όπου είχε συμβάλει πάρα πολύ για τη σύνταξή του και η ε, κυρία Γκρέσλε. Ισχύει από 1η Αυγούστου ο κανονισμό αυτό, ε, τρέχοντο, και ήρθε η στιγμή αυτο τρεχοντο εφαρμοστεί η διάταξη του 15.3. Η έρευνα είναι ένα σκέλο σημαντικότατο για την προετοιμασία του μέλλοντο των Ευρωπαίων και του μέλλοντο τη Υπηρού μας. Εδώ όμω δεν καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο ω προ το σημείο αυτό <clears throat> και αναγκαστήκαμε απλώς να ε, διαπιστώσουμε ότι υπάρχει αποτυχία. Από τον Ιανουάριο δεν ξέρουμε κατά πόσο θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε τα 12 τιμόρια. Αλλά θα φανεί από το τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την, το σεβασμό της οροφής του 1% του ΑΕΠ. Ε, και μια νέα πρόταση που ο Επίτροπος Τιγκέρ έχει παρουσιάσει από την Παρασκευή το μεσημέρι. Θα μας την εκθέσει τώρα. Τον ευχαριστώ λοιπόν πολύ που ήρθε και πάλι σας ευχαριστώ κύριε Έτιγκερ για την αφοσίωσή σας και τις άοκνες προσπάθειές σας για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Έχετε το λόγο. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε Αρτουή, κυρίες και κύριοι προβουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε λίγο χρόνο για να σας παρουσιάσω τη νέα μας πρόταση αφού πριν από 11 μέρες δεν επετεύχθη συμφωνία Κοινοβουλίου-Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή, κατόπιν δικής μου προτάσεως, δέχτηκε ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο αύριο θα συζητηθεί στον τριμερή διάλογο. Έχουμε μια σχετική πίεση χρόνου. Αν θέλουμε να προλάβουμε τη σύνοδο της Ολομελίας του Στρασβούργου την άλλη εβδομάδα και θεωρηθεί αυτός ο στόχος και ο τερματισμός αυτής της προσπάθειας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα που έχουμε μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα για να καταλήξουμε. Γιατί το να διαιρεθεί ο προϋπολογισμός του 2018 σε 12 τιμόρια θα σημαίνει μεγάλο πρόβλημα ένα παράδειγμα, τρία παραδείγματα. Πρώτον, η δεύτερη δόση Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδεχομένως να ματαιωνόταν γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα από ό,τι αντιστοιχούν σε ένα 12 Δεύτερον, ε, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο δίνουμε τα χρήματα στα κράτη στους αγρότες και επειδή πηγαίνουμε σε ευρωεκλογέ, δεν θα το κατανοούσαν καθόλου. Αλλά επίσης και αυξήσει ε, στα θέματα της έρευνας ε, θα ε, ήταν ενδεχομένω αναγκασμένες να ματαιωθούν και κάποια άλλα προγράμματα που μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε δεν θα ήμασταν σε θέση να το πράξουμε. Στη συνδιαλλαγή έχουμε κάνει βήματα πρόοδου, μεγάλα από κοινού και τελικά ένα ή δύο ήταν τα σημεία ε, που ανέτρεψαν τη συμφωνία και μάλιστα η συζήτηση ήταν μέχρι αργά το βράδυ. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες να συμφωνήσουμε αρχαίος, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλησιάζει όσο γίνεται περισσότερο στο όριο των όσων μπορούν να δεχθούν και οι δύο πλευρές. Και μετά από κάποια θέματα που ακούσαμε ότι ήταν σημαντικά για το Συμβούλιο και άλλα για το Κοινοβούλιο, καταρτήσαμε αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού. Παραμένουν τα κέντρα βάρος, ε, αποτελεσματικότητα, ανάπτυξη, χρήματα για τη μετανάστευση, την πολιτική ασφαλείας και αύξηση ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής. Έρχομαι στην διαφάνεια υπαριθμό 3. Η ανάληψη υποχρεώσεων αντιστοιχεί στο 1,00 ε, του ΑΕΠ. 165,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018, αυτό ε, συνιστά αύξηση 3,0% για απρόβλεπτες δαπάνες έχουμε ένα περιθώριο 1,3 δισεκατομμύρια που κατά την άποψή μας είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Για τις πληρωμές τώρα προτείναμε 148,2 δισεκατομμύρια και είναι αύξηση κατά 2,4% σε σχέση με τον προπολογισμό του περασμένου έτους. Έχουμε στην τέταρτη διαφάνεια. Με εξαίρεση το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ΕΦΣΥ, στον τίτλο 1α έχουμε αυξήσει τα κονδύλια κατά 3 δις περίπου. Για τον ορίζοντα 2020 προτείνουμε και άλλη αύξηση 100 εκατομμυρίων, μια επιπλέον αύξηση και μάλιστα βάσει του άρθρου 15.3. Δηλαδή, συνειδητά δεν έχουμε προσθέσει 400 εκατομμύρια, αλλά 100. Και αυτό είναι μια χειρονομία καλή θέληση ότι δεν θέλουμε να συγκρουστούμε, αλλά λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά τι επιφυλάξει του Συμβουλίου. Επανέρχομαι στα 400 εκατομμύρια. Αυτά προέρχονται από το 2017, αλλά όχι αποκλειστικά από το οικονομικό έτος 2017. Αλλά το 2017, από το έβδομο ερευνητικό πρόγραμμα, το προηγούμενο δηλαδή, του προηγουμένου ε, δημοσιονομικού πλαισίου, μεσοπρόθεσμου, ε, έγινε η εκαθάριση δηλαδή για την προγραμματική περίοδο 2007 με 2013, εγγράφησαν στον προϋπολογισμό αναπορόφητα κονδύλια, συν τα αναπορόφητα του 2017. Εξού και το υψηλό ποσό αυτό, 400 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 100 θέλουμε να τα εγγράψουμε ως νέα εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2019. Για το έρασμος συν θέλουμε αύξηση της τάξης των 200 εκατομμυρίων Ε, και συνολικά είναι 400 εκατομμύρια επιπλέον για το 2019 σε σχέση με το 2018 για το Erasmus. Στο κόσμο έχουμε μια μικρή αύξηση και στα άλλα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 5 εκατομμύρια ευρώ. Αν κοιτάξετε και πάλι και θέλετε να μελετήσετε το άρθρο 15.3, θα πρέπει να διαβάσετε τη διαφάνεια υπαριθμών 5. Θα ήθελα εδώ να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Κύριε Πρόεδρε, προηγουμένως αναφερθήκατε ε, στο νέο άρθρο και στην κυρία Γκρέσλε που ήταν αρμόδια εισηγήτρια για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και διαπραγματεύτηκε το συγκεκριμένο άρθρο 15.3 με το Συμβούλιο ε, ε, το νέο αυτό άρθρο δημιουργεί λοιπόν τη δυνατότητα. Κάποια κονδύλια που δεν έχουν απορροφηθεί γιατί καταργήθηκε η θέση τους να εγγραφούν και πάλι στον προπολογισμό. Ε, εναπόκειται στο Συμβούλιο να το συμφωνήσει με το Κοινοβούλιο. Δεν είναι αυτόματη αυτή η διαδικασία, αλλά δεν σημαίνει ότι καταρχήν είναι απορριπταία είναι μια νέα δυνατότητα ε, που δημιουργείται με το νέο ε, δημοσιονομικό κανονισμό. Και την περασμένη Παρασκευή για πρώτη φορά ε, παρουσιάσαμε τη νέα μας πρόταση στο Συμβούλιο. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής, κύριος Κόπμαν, είναι αρμόδιος και μια σειρά κρατών μελών βλέπουν ουδέτερα αυτή τη χρήση του άρθρου 15.3 και τα 100 εκατομμύρια. Υπάρχουν άλλα κράτη που το επικροτούν και γύρω στα 10 κράτη-μέλη ε, είναι αρνητικά και απορριπτικά στη στάση τους. Και αυτό αύριο σίγουρα θα κυριαρχήσει στις ε, συζητήσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν αποχρόντες λόγοι για αύξηση των κονδυλίων, ιδιαίτερα στην έρευνα και μπορούμε αυτό να το τεκμηριώσουμε και να το αποδείξουμε. Έρχομαι στον τίτλο 1β τώρα, που είναι η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Έχουμε αυξήσει την αρχική μας πρόταση κατά 117 εκατομμύρια και το 2019 έτσι θα έχουμε ακριβώς το ίδιο ποσό με το 2018 για την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Στο τίτλο 2, Γεωργία. Καταπολέμηση της πανόλησης του χείρου της Αφρικανικής και το θέμα του ελαιολάδου. Είναι όλα αυτά τα θέματα που συζητούνται στην συνδιαλλαγή. Για το πρόγραμμα LIFE και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης θέλουμε να αυξήσουμε τα κονδύλια. Και μάλιστα είναι μεγαλύτερη πρόταση από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τώρα στον τίτλο 3. Ασφάλεια και ε, ηθαγένεια και ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Άμεφ, 400 εκατομμύρια. Σημαντική αύξηση για το ταμείο αυτό. Εμείς θέλουμε η αύξηση είναι της τάξης του 65%. Και το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Γκάιερ για την Ιουλίζα, Europol και Eurojust, για τους οργανισμούς αυτούς και για το Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη, ε, Multimedia και άλλα. πολέμηση των ψευδών ειδήσεων, των fake news. Στην κατηγορία, ε, στον τίτλο μάλλον 4, παραμένει μέγα πρόβλημα η χρηματοδότηση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Ε, έχουμε σημειώσει τις επιφυλάξεις του Κοινοβουλίου, τα 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 2 δισεκατομμύρια από τα περιθώρια είναι ένα δις ε, καινούργια. Έχουμε και το μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία και τα διάφορα προγράμματα γειτονίας, 21 εκατομμύρια αύξηση και για τα Ηνωμένα Έθνη επίσης. Για να χρηματοδοτήσουμε λοιπόν τη γειτονία, την αναπτυξιακή βοήθεια και την καταπολέμηση των αιτίων που οθούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση. Αυτό ανταποκρίνεται περίπου ε, στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Επίσης ζητήσατε να μειωθεί η προενταξιακή βοήθεια που δίνεται στην Τουρκία και μάλιστα εμεί δώσαμε συνέχεια σε αυτό, αντιδράσαμε. Στον τίτλο 5 έχουμε την προσαρμογή των υπηρεσιών σε σχέση με την προσαρμογή των μισθών που είναι χαμηλότερη της αναμενόμενης 20 εκατομμύρια και επίσης μείωση των δαπανών για τα κτίρια προτείνουμε μικρές αυξήσεις για το δικαστήριο και για τη στρατηγική επικοινωνία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. όλα τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που πρότεινε το Κοινοβούλιο ε, λήφθησαν υπόψη απολύτως και πλήρως. Έρχομαι τώρα στην 7η διαφάνεια. Εδώ βλέπετε τις αυξήσεις της ανάληψης υποχρεώσεων στο δεύτερο σχέδιο του προπολογισμού και συνολικά οι αυξήσεις αυτές είναι περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ και η μερίδα του Λέοντος είναι τίτλος 1α, 1β και 4. Προτεραιότητες και για το Κοινοβούλιο αυτές. Και πιστεύουμε ότι έχουμε ανταποκριθεί κατάλληλα ε, στις προσδοκίες ε, του Κοινοβουλίου. Όγδοη διαφάνεια. Εδώ έχουμε κάποια ειδικά μέσα που επιτρέπουν ε, να υπερβούμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το αξιοποιούμε. Το μέσο ευελιξίας, ας πούμε, για την ανάληψη υποχρεώσεων και για τις πληρωμές, ε, μπορεί να αξιοποιηθεί και σε ένα ποσό που φτάνει μέχρι τα 2,45 δισεκατομμύρια. Άρα παραμένει για το 2019 ε, ένα ποσό 1,8 δις για απρόβλεπτες δαπάνες και έκτακτες καταστάσεις. Έχουμε λοιπόν περιθώρια για θεομηνίες, ε, καταστροφές και άλλα απρόβλεπτα. στις επόμενες διαφάνειες. Στην 9 ε, είναι το χρονοδιάγραμμα, αύριο συνεδριάζει ο τριμερής διάλογος και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε αύριο να επιτευχθεί συμφωνία και με βάση αυτή τη συμφωνία ε, να έρθει ε, στο Στρασβούργο στις 12 ή στις 13 του μηνός το θέμα για να γίνει συνολική επιτελική ψηφοφορία. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να συνεδριάσει ή θα πρέπει να συνεδριάσει η δική σας Επιτροπή στο Στρασβούργο στι 10 του μηνό για να λάβει τι αποφάσει. τη. Βλέπετε ότι ο χρόνος πιέζει. Να σας πω κάτι για τα προσωρινά 12 τιμόρια. Ε, είναι κάτι το πολύ αρνητικό για ε, τις υποχρεώσεις που έχουμε για το 2019 και θα έχει αρνητικέ επιπτώσει αυτό το σύστημα των 12 τιμωρίων για όλου. Μετανάστευση, γεωργία, ορίζον 2020, Εράσμου ΣΥΝ. Δεν θα μπορούμε να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Κάτι που θα γινόταν αν εγκρινόταν ο υπολογισμό, δηλαδή αυξήσει. Δεν μπορούν να γίνουν με τα 12 τιμόρια αυτέ οι αυξήσει. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Για τη γεωργία οι άμεσες ενισχύσεις ε, στους αγρότες θα πρέπει να καταβληθούν από τα κράτη-μέλη. Αλλά ξέρετε ότι 75 με 80% των πόρων καταβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Με τα 12 τιμόρια δεν γίνεται αυτό. Ε, γιατί αντί για το 75-80% μπορεί να δίνεις κάθε μήνα 8,3% υποθέτω ότι δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει αυτό στους αγρότες. Και στο Erasmus Συν περίπου 400.000 υποτροφίες θα καθυστερήσουν. Τα δύο τρίτα περίπου όλου του προγράμματος ε, καταβάλλονται ή συνδέονται στο πρώτο τρίμηνο. Ένα δωδεκατημόρια, έστω και τρία δωδεκατημόρια δεν φτάνουν σε καμία περίπτωση. Για τον ορίζοντα 2020, πάλι με το σύστημα των 12 τιμωρίων, Ήδη από τον Ιανουάριο ε, λείπουν 100 εκατομμύρια για τις πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Για μισθούς, 2.000 ερευνητές δεν μπορούν να πληρωθούν το μισθό τους. Τέτοιες ε, καταστάσεις δεν μπορεί κανείς να τις επιθυμεί για το ε, Connecting Europe, την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Θα υπήρχε επίση πρόβλημα για το ΣΕΣΑ, για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και διάφορα άλλα προγράμματα. Θα μπορούσα να σας απαριθμώ εδώ ακόμα πολλά ε, προγράμματα και ονόματα προγράμματων. Το νέο hotspot στη Σάμο θα καθυστερήσει να κατασκευαστεί. Ε, ο Frontex επίσης δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί κτλ. κτλ. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να συμφωνήσουν αύριο και οι τρεις πλευρές, Κοινοβούλιο, ε, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήταν ευχής έργο. Και τέλος, ε, έρχομαι στην ενδέκατη διαφάνεια. Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 προβλέπει αυξήσεις για τις δικές σας προτεραιότητες. Επενδύσεις, ε, απασχόληση των νέων, ασφάλεια 5 δις ευρώ, 3,1% είναι η αύξηση. Θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο προπολογισμός του 2019. Ένα στιβαρό, γερό προπολογισμό που να ανταποκρίνεται και στι προσδοκίε μια εκλογική χρονιά. Είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει και η Γενική μου Διεύθυνση και το ιδιαίτερο γραφείο μου και για ε, σήμερα και για αύριο στη διάθεσή σας. Αν θέλετε διευκρινήσεις για αριθμούς, για ποσά, ελάτε, αποταθείτε σε μας πριν το τριμέρι διάλογο, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε τον κοινό χρόνο που θα έχουμε εκεί ε, κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Δηλαδή να έχουν ξεκαθαριστεί τα θέματα αυτά, τα διευκρινιστικά για τα ποσά, πριν πάμε να συναντήσουμε το Συμβούλιο. Για να διαλύσω και οποιασδήποτε αμφιβολίες, για να λύσω απορίες που έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και για την ε, ευκρίνεια αυτής της παρουσίασης. Τώρα, για τις ε, δυσκολίες με το 12 πρέπει να προσθέσουμε και άλλη μια δυνατότητα, τη χρηματοδότηση του δισεκατομμυρίου για την Τουρκία. Και αυτό είναι μία από τις συνέπειες της έλλειψης ε, συμβιβασμού, εάν τελικά αυτό συμβεί. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν ο κ. Τανιλεβιώτη θα έχει το λόγο που είναι ο Γενικό Εισηγητή. και συγχωρήστε με αλλά θα σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε τα έξι λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες που και πέντε λεπτά θα μου έφταναν. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και του συνεργάτε του, την ομάδα των συνεργατών του, διότι εργάστηκαν τόσο ε, επιμελώς και σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες και εννοείται και του προηγούμενου μήνε και αυτές τις προηγούμενε ώρες. Ήμασταν διαρκώς σε άμεση επικοινωνία και με μένα τον ίδιο και με τους υπόλοιπου συναδέλφου και όδους εισηγητές και γενικώ με τα μέλη τη επιτροπή μα. Τι να πω. Την Παρασκευή λάβαμε το έγγραφο και μπορέσαμε να το δούμε και να το μελετήσουμε. Δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα να θέσω στον Επίτροπο. Θα τα συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς και αύριο στην προπαρασκευαστική μεταξύ μας για να καταρτήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Έχω μία μόνη ερώτηση να θέσω στον Επίτροπο. Ακούει το Συμβούλιο σας άκουσε, υπάρχει περίπτωση να δεχτεί αυτή την πρόταση. Διότι δικαίως μας λέτε ότι πρέπει να βιαστούμε. Και κάθε μέρα που περνάει είναι σημαντική. Για να μπορέσουμε όμως να συζητήσουμε και μεταξύ μας και να ξέρουμε τι μας γίνεται και να φτάσουμε στο απόγευμα να έχουμε μια θέση που να μπορεί να οδηγήσει και σε διαπραγματεύσει, πρέπει να γνωρίζουμε λίγο πολύ τι σκέφτεται και το Συμβούλιο για την πρόταση αυτή. Είναι μια πρόταση που κάπω θα μπορούσαν να τη δεχτούν και να τη συζητήσουν ή καθόλου. Για τα 12 τιμόρια, οι προβλέψει που του κάνατε, που μα παρουσιάσετε μόλι τώρα. Του τα είπατε έτσι και στου ίδιου. Και το Συμβούλιο είναι έτοιμο όπω και εμεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Την ευθύνη που εμεί είμαστε σε κάθε περίπτωση πρόθυμοι να αναλάβουμε. Και για την ερώτηση αυτή, ε, Επίτροπε, εσείς καλά κάνατε και μας φέρατε αντιμέτωπους με τις ευθύνε που θα είχε η εναλλακτική να πάμε στην κατεύθυνση των 12 τιμωρίων. Αλλά η απειλή των 12 τιμωρίων δεν μπορεί να είναι ένα μοχλός πίεσης για να αποφασίσουμε ούτε μπορεί να είναι και το κλειδί για να ξεκλειδώσει μια τελική απόφαση από πλευρά μα. Διότι ο φόβο για τα 12 τιμόρια ε, και το τι θα γίνει από το Γενάρη, μιλάμε για μια δεκαπενθήμερη καθυστέρηση. Δεν είναι και κάτι συγκλονιστικό. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι αυτό ο φόβο αυτό των 12 τιμωρίων αυτό που θα κινήσει την Επιτροπή. Το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι αυτό που θα πρέπει να φοβάται να πάει στα 12 τιμόρια. Εγώ το συζήτησα με τους συναδέλφους, επίτροπε. Μάλλον δεν το, δεν το έχω συζητήσει ακόμα με τους συναδέλφους, γι' αυτό και αναλαμβάνω την ευθύνη ενώπιόν τους για, το, για τα λόγια μου. Αλλά για την πρότασή σας, επίτροπε, Εσεί έχετε καμιά ιδέα για το αν Συμβούλιο θα μπορούσε να δεχτεί την πρόταση αυτή, γιατί βάσει τη δική σα απάντηση μπορούμε και εμεί να κάνουμε ήρεμα και συγκροτημένα τι δικέ μα συζητήσει για να φτάσουμε στο απόγευμα με μια θέση έστω και βιαστική και να μπορέσουν επιτέλου να ολοκληρωθούν ενδεχομένω οι διπλωματεύσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε κύριε Γενική Συγητά. Ο κύριο Γκάγερ. Για του οργανισμού, Δεν έχει να πει τίποτα. Ο Πάλου Ρεμπίχ τίποτα. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στους σκιώδεις που θα ήθελα να μην μιλήσουν για πάνω από τρία λεπτά ο καθένας και βέβαια η Μόνικα Όλμαγερ είναι η πρώτη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, παρουσίαση και την πρόοδο με βάση τα όσα ε, συζητήσαμε στο παρελθόν. Και χαίρομαι και για το 15-3 το οποίο τον προσφέρεται ως κλάδον ελέας. Ε, υπό ποια έννοια. Ότι δεν θέλουμε τα 400 εκατομμύρια και την πλήρη συμπεριλήψη, αλλά ότι το 15-3 δεν είναι ένα ε, όπλο το οποίο... Ε, αποκλείεται, παραγωνίζεται και πριν γεννηθεί ακόμα ε, καθίσταται ξεπερασμένο. Το Συμβούλιο πώς θα τη δράσει αυτό. Γιατί θεωρώ ότι ορισμένοι οικονομικοί υπάλληλοι δεν θα ήθελαν ποτέ να προκύψει ε, αυτό το άρθρο 15.3 γιατί μπορεί να διακηρύσουν διάφορα εκατομμύρια και να τα μοιράζουν αλλά όταν καλούνται να τα υλοποιήσουν θα προτιμούσαν να μην το κάνουν. Επίση, θεωρώ θετικό την αύξηση του ορίζον 2020 και των ερευνητικών ε, πόρων. Για το κόσμο ε, είναι μικρή αύξηση. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πίεση που υφίσταται το πρόγραμμα αυτό. Είναι από τα προγράμματα που πιέζονται πολύ. Για την ΕΑΣΟ η νομοθεσία έχει εξαιρεθεί. Κάτι που το θεωρούσαμε εμείς δεδομένο τώρα δεν το έχουν βγάλει και θεωρούν ότι θα λυθεί ε, με διορθωτικό και συμπληρωματικό προϋπολογισμό όταν εγκριθεί ο λόγο κανονισμός. Τα ίδια για την ΕΣΜΑ, για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, EBA, τις διάφορες εποπτικές αρχές. Ε, επίσης θεωρώ πολύ θετικό τουλάχιστον ότι δεν βγήκανε τα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί ειλικρινά Πώς μπορεί κανείς να θέλει στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια όταν το Ταμείο είναι μείον. Θα ήταν μεγάλη δυσκολία. Ειλικρινά. Και στο είπα το πρωταξικό για την Τουρκία, εγώ θα έκοβα ακόμα περισσότερα, γιατί αν δούμε τι κάνει και το Συμβούλιο και τι προτείνει, εντάξει θα δείξει. Ε, γενικά, ως αφετηρία, είναι πολύ καλή η πρόταση αυτή. Γιατί ερχόμαστε πιο κοντά στη θέση του Κοινοβουλίου και στα όσα είχαμε ζητήσει από πέρσι Κάτι που θέλω να ρωτήσω τον Επίτροπο για το τίτλο 5 που με προβληματίζει ακόμα. Θυμάμαι στη συνδιαλλαγή ότι η Αυστριακή Προεδρία επαναλάμβανε ότι πρέπει να γίνουν περικοπές στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει το 5%. Το τηρήσαμε το 5%. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάπως αφόρητα. Έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι τώρα προσπαθούν ε, να αφεμάξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά της και να ενισχύσουν την κυριαρχία του Συμβουλίου. Και αν πέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, έχει ε, απόθεμα και εφεδριές με τους υπαλλήλους των διαφόρων Υπουργείων στα κράτη-μέλη. Εμείς αυτά δεν τα διαθέτουμε ως πόρους ε, ανθρώπινους. Θα ήθελα να το πω και να το τονίσω ότι για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση αυτή από πλευράς του ΕΛΚ να τη δεχτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Κέλμελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε Οτιγκερ, σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την δουλειά αυτή, την εμπεριστατωμένη και την πρόταση που έχετε εκπονήσει με το επιτελείο σας και με τον τρόπο το πολύ ευσύνοπτο που μας παρουσιάσετε αυτά τα θέματα σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλό ως αφετηρία για να προχωρήσουμε. Τώρα δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα επιχειρήματα που έχουμε εμείς ως πολιτική ομάδα κατά της ε, πρότασης του σχεδίου του προπολογισμού παραμένουν, τα έχετε ακούσει, τα έχουμε παρουσιάσει, αλλά τελικά θα πρέπει να δεχτούμε ότι όταν υπάρχει μια πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο για μια συγκεκριμένη διαδικασία, τι να κάνουμε, έχει αποφασιστεί δημοκρατικά. Θα το δεχτούμε. Ε, κάπου που έχουμε αντιρρήσεις, είναι στη χρήση και εφαρμογή του άρθρου 15.3 για λόγους διαρθρωτικούς και ε, αρχής όντως αυτό το μέσο δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί με τον τρόπο που το προτείνεται. Ακόμα και αν πρόκειται μόνο για 100 εκατομμύρια εντό εισαγωγικών, είναι θέμα αρχής, όπως και με τους ιδίους πόρους. Είτε τους θέλουμε, είτε δεν τους θέλουμε. Εάν τους έχουμε, έστω και με ομοιοπεθετικά ποσά, ε, πολύ γρήγορα θα έρθουμε αντιμέτωποι ε, με το γεγονό ότι θα πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο και θα παγιώνεται μια κατάσταση. Σας λέω ότι είναι θέμα αρχές. Για τα ποσά νομίζω ότι υπάρχει ε, μια συνένεση, γίνονται βήματα προς την κατεύθυνσή μας και μπορούμε να τα δεχτούμε. Για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και στο Συμβούλιο αυτό το σχέδιο προϋπολογισμού, στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Πρωτοβουλία και τη Χρηματοδότηση, Ενδεχομένω, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε το εξή. Θα μπορούσαμε να φτιάχνουμε αεροπλάνα που να πετάνε οι ηγέτες μας μέχρι την Νότια Αμερική. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον για ορισμένους ηγέτες και ηγέτιδες ε, στην Ευρώπη. Το 15.3 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο αυτό, γιατί έχει να κάνει μόνο με την έρευνα. Νομίζω ότι αυτό περιγράφεται πάρα πολύ ε, λεπτομερώς και αναφέρεται μόνο στην έρευνα. Ζεράρντε Euh, je ne sais pas. Ε, ε, excusez-moi, Monsieur le Président. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, δεν ήθελα να προκαλέσω πρόβλημα και είχαμε κάποιο τεχνικό θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα συνταχθώ κι εγώ με τους ε, συναδέλφους που χαιρετίζουν τις προσπάθειες που κάνουμε, που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη νέα αυτή πρόταση. Πριν λοιπόν να δούμε το θέμα επί της αρχής, Εάν κοιτάξω σφαιρικά τα όσα προβλέπονται για κάποιες από τις δικές μας προτεραιότητες ως ομάδα, δηλαδή την αύξηση 9% για το Horizon 2020 και το 18% για το Erasmus Plus ως αύξηση, όπως μια μικρότερη αύξηση για το κόσμο και θα μπορούσα να συνεχίσω να πω γενικά για το σύνολο των προτεραιοτήτων της ομάδας μου έχουμε ε, αρκετή αύξηση στην, ε, στα ποσά αυτά που μπορούν να μας ικανοποιήσουν. Όμως είναι πολύ λίγα τα μέσα τα οποία θα κινητοποιηθούν για να δώσουμε τη μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος. Και το λέω ε, αυτό γιατί χτες έγινε και μια μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες πιέζοντας το να αυξηθούν τα χρήματα που διαθέτουμε. Έχω λοιπόν εκεί κάποιες επιφυλάξεις και επιφυλάξεις για τα σχόλια τα οποία ζητήσαμε να συμπληρωθούν και δεν είναι εδώ. Αλλά ο συνάδελφος Βιωτήκ είμαι σίγουρος πως θα τα ε, ξαναβάλει στο τραπέζι διαπραγμάτευση παρόλο που βλέπω ότι δεν με ακούει εδώ. Παντώ θα του μιλήσω σε λίγο για να το κάνουμε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα το οποίο δεν λύνεται. Γιατί στις διαπραγματεύσεις αυτές έχουμε καταρχήν το θέμα της ουσίας και του περιεχομένου του προϋπολογισμού αφενός και πιστεύω πως η προσπάθεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια εξαιρετική βάση από τις οποίες μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις. Ως βάση συζητήσεων μόνο στηρίζουμε αυτή την πρόταση. Αλλά έχουμε και το αφετέρου που είναι ένα θέμα θεσμικής τάξης. Η συνθήκη προβλέπει να έχουμε δύο δημοσιονομικές αρχές. Δύο βραχίονες που θα πρέπει να διαπραγματεύονται για να καταλήξουν σε συμφωνία. Το Συμβούλιο μας είπε για την ε, Τουρκία πως εκεί δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση. Μας είπαν δεν θα το συζητήσουμε καθόλου, ό,τι προτείνουμε θα το ε, δεχτείτε, αλλιώς δεν υπάρχει κοντήλη στον προϋπολογισμό. Και εμείς, εμείς λέμε το 15-3, εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Και γιατί το βρίσκουμε ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί έχει να κάνει με κονδύλια για τα οποία ήδη στο παρελθόν υπήρξε συμφωνία, συμφωνία και για την ανάληψη της δέσμευσης αλλά και για την δαπάνη, την εκτέλεση της δαπάνης. Και δεύτερον, γιατί ο μηχανισμός ο οποίος είχε στηθεί από τον ε, χρηματικό κανονισμό είχε πει πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον κλάδο της έρευνας. Δεν μιλώ για το ύψος του ποσού. Προτιμώ το σύνολο των κονδυλίων να φτάσει αυτά τα 400 συν εκατομμύρια. Αλλά αν έχουμε το 15.3 εδώ στη διάθεσή μας, θα μπορούσα να συμφωνήσω με κάποιες μικροποσαρμογές επ' αυτής της πρότασης. Αν όμως δεν το έχουμε, εγώ δεν θα πάω στην ομάδα μου και να υποστηρίξετε τούτο το προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν κλείσαμε και με τους σκιώδες ομιλητές που είναι παρόντες. Τώρα, οι σκιώδες για τα υπόλοιπα. Κυρία Κόλμελ για τα υπόλοιπα τμήματα. Κυρία μου, δεν σας είχα δει. Ευχαριστώ πολύ. Με βάλαν στη γωνία για να μην ε, συμπεριφερθώ, γιατί φαντάζομαι συμπεριφερθήκα άσχημα σε κάποια προηγούμενη συνάντηση και γι' αυτό με κρύψανε. Εν πάση περιπτώσει, πολλά είχαμε να πούμε και τις περασμένες φορές και για το 5 γιατί εκεί έχουμε κάποιες τροποποιήσεις ε, που μας επιτρέπουν να μειώσουμε το ύψος της πρότασης και αυτό μας βοηθά στο να τετραγωνίσουμε καλύτερα τα στοιχεία. Επειδή έχω το λόγο, για να μην τα πω και πάλι, θα κάνω όλα μου τα σχόλια. Καταρχήν θα ήθελα να κατανοήσουμε όλοι τι έγινε στην τελευταία συνδιαλλαγή είχαμε λάβει μία πρόταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, η οποία σε γενικές γραμμές ήταν παρόμοια με αυτή που έχουμε τώρα, με κάποιες προσαρμογές στα αριθμητικά στοιχεία. Όμως, φύγαμε γιατί το Συμβούλιο δεν δεχόταν τι γενικές γραμμές αυτής τη πρόταση, δεν δεχόταν πουδενή το 15-3 και επιπλέον στα αριθμητικά στοιχεία και στα νούμερα ήθελε και άλλες περικοπές. Εκεί λάβαμε την απόφαση. Δεν φύγαμε επειδή το επιθυμούσαμε. Φύγαμε γιατί η πρόταση που είχαμε πάνω στο τραπέζι δεν επρόκειτο να τύχει διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο. Όχι γιατί δεν ήταν ιδανική. Άρα λοιπόν, το είπε ο εισηγητής, το είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, το επαναλαμβάνω και εγώ. Το Συμβούλιο, τι λέει. Γιατί αν μπορεί τη γενική φιλοσοφία να τη δεχτεί, να μπούμε και στις λεπτομέρειες ανά αν δεν μπορεί, θα επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση στην οποία, ε, την οποία αντιμετωπίσαμε την τελευταία μέρα της συνδιαλλαγής. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν και πάλι το εξή. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε 12 τιμόρια προσωρινά. Ξέρουμε τι προβλήματα δημιουργούν. Όμως, δεν πρόκειται επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό να δεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση μας κατεβάσουν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε τι πιστεύει το Συμβούλιο για να δούμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, να δώσουμε εντολή στον εισηγητή μας για να διαπραγματευτεί τις λεπτομέρειες, να δούμε αν υπάρχει περιθώριο προσαρμογής των προτάσεων και στο επίπεδο των αριθμών. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αν έχουν γίνει δεκτές αυτές τις προτάσεις επί της αρχής ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κολμέλ. Όχι. Εσείς είχατε σχολιάσει και το 3 και όλα τα υπόλοιπα μαζί. Οπότε, κύριοι συνάδελφοι, εκτός από τους σκιάδες, ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση αυτή. Θα ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Θα σας ευχαριστήσω για τη δουλειά που κάνετε γιατί είσαστε πραγματικά, κάνετε ποιοτική δουλειά, πολύ επαγγελματική και μάλιστα με μεγάλη πίστη σε αυτό που είμαστε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Κανείς, μα κανείς δεν θα μας καταλάβει αν ξεκινήσουμε το 2019 με προσωρινά 12 τιμόρια. Γιατί τι έχουμε στο τραπέζι. 0,9 χάνεται το μικρόφωνο το μεγαλύτερο, με συγχωρείτε, του ΑΕΠ μας είναι ε, στο τραπέζι του διαπραγματεύσεων. Είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά ιστορικά. Κανείς πολίτης, Γερμανός, Γάλλος, δεν θα μπορέσει να κατανοήσει γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη ευνοούμενη από την έρευνα, ε, να μας πούνε, μα εσείς ευνοείστε από την έρευνα και δεν θέλετε να την ενισχύσετε. Έχετε λάβει δεσμεύσεις και δεν τις έχετε φέρει σε πέρας. Και τώρα δεν μιλάμε καν για αυτές τις ε, δεσμεύσεις. Μιλάμε 100 εκατομμύρια ευρώ. Και ο μεγαλύτερος, η χώρα που έχει πιο πολύ ευνοηθεί είναι η Γερμανία και η τρίτη χώρα από τις πιο ευνοούμενες είναι η Γαλλία. Αυτά τα λέω και θα κλείσω λέγοντας πως ίσως ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας θέλει να ξεκινήσουμε με τα προσωρινά δωδεκατημόρια. Μπορεί να το επιθυμεί και ο Υπουργό Γάλλος Οικονομικών, αλλά είμαι σίγουρος πως η καγκελάριος κυρία Μέρκελ δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και ούτε ο πρόεδρος Μακρόν. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε στο επόμενο πολιτικό επίπεδο, γιατί η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή, Ένω... στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασταθής. Και αν υπάρχουν υπουργοί οικονομικών που θέλουν αυτή την αστάθεια να την ενισχύσουν ή να την προωθήσουν, το λέω δημόσια, θα πρέπει να το πούν ανοιχτά. Εμείς αυτό που επιθυμούμε πάντα είναι το καλύτερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη σταθερότητα. Και ένα προπολογισμό ο οποίο θα είναι ρεαλιστικός, και παράλληλα θα είναι και υπεύθυνο. Ευχαριστούμε ο κύριος Μουρεσάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να ευχαριστήσω τον Επιτροπό Έτιγκερ για αυτή την πρόταση του δεύτερου σχεδίου προπολογισμού και που ήρθε προσωπικό να μα την παρουσιάσει. Το πρώτο που θέλω να πω είναι το εξή. Αποτύχαμε στην πρώτη μα απόπειρα, και αυτό δεν ήταν καλό για την αξιοπιστία όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ούτε για το Συμβούλιο, ούτε για την Επιτροπή, ούτε για εμά εδώ στο Κοινοβούλιο. Και το είδαμε ήδη να αναφέρεται και στον τύπο αυτό. Αλλά ας είμαστε ειλικρινεί. Δεν ήταν και δράμα ότι δεν συμφωνήσαμε στην πρώτη προσπάθεια. Όμω θα είναι δράμα τη δεύτερη φορά και αρκετά τραγικό ε, αν δεν συμφωνήσουμε τη δεύτερη. Θα είναι πολύ κακό για την αξιοπιστία τη Ένωση, θα είναι πολύ κακό για τα κράτη-μέλη και θα είναι κακό και για του δικαιούχου. Ε, κατά κύριο λόγο, όπω είπε και ο Επίτροπο. Ε, απλώς να επισημάνω ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και ότι είναι πολύ δύσκολες οι διπλωματεύσεις αλλά αυτό δεν αρκεί, διότι αντίξωες συνθήκες και εκπλήρωση των υπεχρεώσεων τους έχουν εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πυροσβέστες, ε, τραυματιοφορείς, ε, γιατροί, νοσοκόμες, όλοι εργάζονται υπό αντίξωες συνθήκες και τα καταφέρνουν. Άρα και εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε τη δουλειά μας και να φέρουμε ένα προπολογισμό στο τραπέζι πριν τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό, Ντανιέλε, πιστεύω ότι πρέπει να δείξουμε πυγμή στι διαπραγματεύσει. Πρέπει να ορίσουμε με αυστηρότητα κάποια, κάποιες, κάποια όρια, κάποια απαγορευτικά όρια και κόκκινε γραμμέ. Πρέπει να γίνουν σεβαστά αυτά, αλλά πρέπει να είμαστε και επικοδομητικοί. Πρέπει να επιζητήσουμε λύσει και να βρούμε απαντήσει στι προτάσει του Συμβουλίου. Πρέπει να, θε, να ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο, ακριβώ όπω εξήγησε μόλι τώρα ο Ζωζέ Μανουέλ Φερνάντε. Η δική μου λοιπόν η γραμμή είναι να ορίσουμε τι κόκκι, απαγορευτικά μα όρια, αλλά να είμαστε και επικοδομητικοί. Να είμαστε έτοιμοι να εξεύρουμε λύσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι βήμα-βήμα θα πάμε τελικά σε αυτό που λέει από την αρχή το Συμβούλιο που έχει μείνει μετακίνητο στη θέση του. Πιστεύω το σχέδιο προπολογισμού που έχει υποβάλει η Επιτροπή είναι πολύ καλό σημείο αφετηρία για να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τι διαφορέ μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Οι διαφορέ αυτέ είναι προφανώ επαρκτέ, ιδάλω δεν θα είχαμε αποτύχει όμως οι προτεραιότητές μας ε, είναι σίγουρα προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση, αλλά να εργαστούμε για το σχέδιο προπολογισμού, ασκώντα κάθε δυνατή πίεση. Διότι στο τέλο, ε, στο κάτω-κάτω τη γραφή, αυτό που θέλουμε είναι ένα προπολογισμό στον οποίο έχουμε συνεισφέρει, αλλά δεν μπορούμε να τον εγκρίνουμε και μόνοι μα μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί το Συμβούλιο. Πρέπει να είμαστε οικοδομητικοί και με αυτού. Ευχαριστούμε. Κανεί άλλο δεν ζητά το λόγο από ό,τι βλέπω. Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ τη δική μου προσωπική άποψη. Ε, να υπογραμμίσω ξανά ότι είναι ο τελευταίος μας προπολογισμός, ο τελευταίος προπολογισμός αυτής της θητείας. Πρόκειται για μια μέγιστη σημασίας πολιτική πράξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φρονώ, ε, υποβάλλει μια πρόταση που για μας ε, είναι η ελάχιστη που θα μπορούσαμε να αποδεχτούμε. Διότι εάν έπρεπε να απαρνηθούμε ε, τις προτεραιότητές μας, τι εικόνα θα έδινε το πολιτές δημοσιονομικό μας πλαίσιο 2021-2027 με μια τέτοια λογική και πνεύμα. Θα ήθελα λοιπόν αύριο το απόγευμα στον τριμερή διάλογο να προχωρήσουμε με τρόπο θετικό και ξαναυπόθηκε επανειλημμένω και στη διάρκεια τη Ανδιαλλαγή. έχουμε πολλέ φορέ την αίσθηση ότι από τη μια είναι το Κοινοβούλιο, από την άλλη το Συμβούλιο, αλλά το Συμβούλιο πολύ συχνά ε, εκπροσωπείται από του υπαλλήλου των Υπουργείων Οικονομικών που ε, τοποθετούνται. Αλλά δεν υπάρχει πολιτική πυγμή, δεν υπάρχει κρατική εκπροσώπηση, δεν υπάρχει κάποιο από την κυβέρνηση. Αυτοί φαίνεται σαν να μην αδιαφορούν. άρα πρέπει να υπάρξει και κάποια πολιτική ανάληψη ευθύνη. Μπορεί αυτή να εκφραστεί είτε εδώ είτε με άλλο τρόπο αλλού. Ε, βλέπουμε όμως την οργή των πολιτών. Είναι ε, δυσαρεστημένοι με την διαχείριση των κρατικών πραγμάτων από, την από τις κυβερνήσεις. Έχουν την αίσθηση ότι την εξουσία έχουν καταλάβει τεχνοκράτες. Εδώ λοιπόν η έρευνα ω συμβιβαστική λύση στον προπολογισμό του 2019 θα πρέπει να προβάλλει πάνω απ' όλα το πολιτικό μα όραμα και όχι την τεχνοκρατική προσέγγιση. Ε, έχω να αποθέσει τι ελπίδε μου στι ώρε που βρίσκονται μπροστά μα μέχρι αύριο το απόγευμα και καθένα από εσά, συνάδελφοι, κυρία Γενική Εισηγητά, υπεύθυνη για του οργανισμού, εισηγητέ για, τα υπόλοιπα τμήματα του προλογισμού και εσεί, Επίτροπε, Ελπίζω να μεταφράσετε τις προσωπικές απεπιθήσεις και την ε, ικανότητά σας ε, να πείσετε ε, να το καταφέρετε και να έρθει κάποιο θετικό αποτέλεσμα αύριο στο Κορεπέρ. Ο κύριος Βόν έχει ζητήσει το λόγο. Ακούω. Βασίζω λοιπόν τις ελπίδες μου στο αυριανό απόγευμα, ίσως βράδυ, ίσως και μέσα στη νύχτα, ίσως ξημέρωμα της Τετάρτης. Κύριε Επίτροπε, ποια είναι η δική σας η άποψη στο τέλος αυτής της συζήτησης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την, κατά τη γνώμη μου, πάρα πολύ επικοδομητική συνεισφορά σας με τις παρεμβάσεις σας. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή σας. Με ρώτησε ο κύριος Βιώτη τι φρονεί το Συμβούλιο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ο κύριος Γενικός Διευθυντής σήμερα το μεσημέρι ε, παρουσίασε τη νέα μας πρόταση στο Συμβούλιο και έγινε και μια πρώτη συζήτηση σχετικά. Η οποία αφορούσε κυρίως τα ποσά, το ύψος του προπολογισμού, γιατί υπάρχουν ακόμα φωνές που δεν είναι ικανοποιημένες με την αύξηση που προτείνουμε. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη πολύ επικριτικά για το άρθρο 15.3. Κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν θέλουν καν να εφαρμοστεί αυτό το άρθρο. Κατά τα άλλα όμως είμαστε θετικοί και θέλουμε την πρότασή μας να την δώσουμε ως αφετηρία ε, για τη συζήτηση και αυτό δεν το απορρίπτει το Συμβούλιο, το δέχεται. Κυρία Χολμάγερ, το βλέπω όπως και εσείς. Οι ε, περικοπές σε προσωπικό ε, δεν είναι σκόπιμες ούτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε πουθενά άλλο. Ε, έγιναν οι περικοπές του 5% και όταν αποφασίστηκε αυτό το 2013 ε, υπήρχε και κάτι άλλο που αποφασίστηκε ότι το 2022 θα υπάρχει μια ισορροπία, μια σταθερότητα. Αυτά θα ε, συζητηθούν στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αλλά όχι για τον προπολογισμό του 19, ούτε του 20 άλλωστε. Δεν αλλάζει αυτό. Και έχω περίπου αντίστοιχη αντίληψη με εσάς, κυρία Χολμάγερ. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μόνο τους υπαλλήλου του. Ε, το Συμβούλιο δεν έχει μόνο τους υπαλλήλου εδώ του Συμβουλίου, αλλά και τους ε, υπαλλήλου των Υπουργείων στα κράτη-μέλη, που μπορεί με ευελιξία να τους χρησιμοποιεί και να τους αξιοποιεί. Το ε, άρθρο 15.3, κύριε Κιόλμελ, είπατε ότι είναι θέμα αρχής. Το σημειώνω αυτό, απλώς θέλω να σας πω το εξής. Επειδή το άρθρο 15.3 προτείνεται μόνο για ε, την έρευνα για το Horizon 2020 και για την Ευρατόμ και σε καμία περίπτωση για άλλο πρόγραμμα αυτή η ε, εφάπαξ ε, εφαρμογή του άρθρου δεν σημαίνει ότι ανοίγει την πόρτα για πάντο επιστητών και για οτιδήποτε. Ειδικά για την έρευνα μπορούν να μεταφέρονται ποσά από ένα οικονομικό έτος στο άλλο, αλλά γι' αυτό πάντα χρειάζεται συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι δεν είναι ευκαταφρόνητη αυτή η σχετική ευελιξία, γιατί υπάρχουν κάποια ερευνητικά προγράμματα που έχουν νόημα και δεν φτάνουν τα κονδύλια. Ενώ υπάρχουν κάποια άλλα κονδύλια που έχουν εγκριθεί για την έρευνα. Δεν έχει νόημα να επιστραφούν και να ψάχνουμε καινούργια χρήματα. Με μεταφορές πιστώσεων εξυπηρετείται ο ίδιος ε, ευγενής στόχος. Και θεωρώ ότι και στο μέλλον ε, σε ένα όγκο, ένα ποσό 11-12 δισεκατομμύρια ε, ή 16 ή 17 δεν θα γαλάσει ο κόσμος αν υπάρχουν μερικά εκατομμύρια ε, που περισσεύουν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος. Αυτό μπορεί να είναι ένα χιλιοστό ε, του συνόλου του ε, προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το άρθρο 15.3 νομίζω είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ ότι είναι μόνο για την έρευνα η εφαρμογή του, όπως άλλωστε προτείνεται κιόλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κατά τα άλλα στη διάθεσή σας και σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημέρι και για σας και για τους βοηθούς σας, τους συνεργάτες σας, κατά τα άλλα ραντεβού στον τριμερή διάλογο. Merci, Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ίσως ο Γενικός Εισηγητής Βιώτη να ήθελε κάτι να πει για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι, ευχαριστώ τον Επίτροπο και φυσικά τις και τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Ο συνήθως ε, ήταν σημαντικές οι συνεισφορές τους. Επίτροπε, πραγματικά το ακούσατε και από τα σχόλια των συναδέλφων. Είμαστε στα τελευταία στάδια της διαδικασίας. Τώρα καλούμαστε, προς στιγμή τουλάχιστον, πώς να το πω, να κάνουμε και μια, ε, ε, έναν απολογισμό του τι κάναμε ως Επιτροπή Προλογισμών ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους τελευταίους μήνες. Είναι ένας απολογισμός για να δούμε και Επίση, κατά πόσον υποχωρήσαμε σε κάποια αιτήματα του Συμβουλίου του τελευταίου ε, μήνε. Δεν είναι μια περίτη διαδικασία αυτοκολακία για να θυμίζουμε στου εαυτού μα πώ συζητήσαμε τον αυτόματο χαρακτήρα κάποιων διατάξεων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο για το άρθρο 15.3, ότι ε, χρειάστηκε να αναχαιτήσουμε τις επανειλημμένες ε, περικοπές που ζητήθηκαν σε πολλές εκδοχές του σχεδίου προπολογισμού. Τις είδαμε, κάποιες από αυτές τις ε, αποδεχτήκαμε, καταλάβαμε τους περιορισμούς του Συμβουλίου δεν ασκήσαμε ουδέποτε ιδιαίτερη πίεση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να κλείσουμε την συζήτηση αυτή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που έκλεισε το θέμα και την παρέμβασή του και ο πρόεδρος Σαρτουή. Δηλαδή χρειάζονται και οι δύο ε, πλευρές, οι δύο διαστάσεις του υπολογισμού. Δηλαδή, εδώ, εάν υπάρχει μία διελκυστίνδα εξουσίας, στην οποία δεν θέλουμε να συμμετέχουμε, που ένας από τους δύο θα κοιτάει αν θα κερδίσει και θα βγει πρώτος, θα βγει ε, ζημιωμένη η Ευρώπη. Ε, ίσως να έχουμε ένα μήνα απουσία έγκρισης του προπολογισμού. Αυτό θα γίνει αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια μονομαχία μεταξύ δύο δυνάμεων που κάποιο θα προσπαθήσει να βγει νικητή. Πρόεδρο, ευχαριστούμε κύριε Γενική Συγητά. Ξέρω ότι η Επιτροπή, ε, ξέρετε κύριε Επίτροπε, ότι η Επιτροπή Κόντε σας περιμένει. Καλή σας τύχη λοιπόν στην παρουσίασή σας αύριο στο Κορεπέρ. Αύριο θα τα πούμε στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστούμε. Την αδελφή τώρα να δώσω το λόγο. Στον κύριο Ashworth, αλλά επειδή δεν έχει έρθει ο κύριος Ashworth, αντικαθίσταται από τον κύριο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι τάχιστος. Θέλω να παρουσιάσω τις μεταφορές. Μεταφορές που έχουν σεβαστεί όλους τους κανόνες και διατάξεις των δημοσιονομικών κανονισμών. Εδώ μιλάμε για ένα έμβασμα που θέλει να ενισχύσει την γραμμή 2001 για την επέκταση και την ανακαίνιση του κτηρίου Κόραντ Αντενάουερ στο Λουξεμβούργο. Μια απόφαση που είχε ήδη ληφθεί ε, από την Επιτροπή Προπολογισμού στις 11 Ιουλίου 2006. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε για τις προτάσεις που μόλις υπέβαλε ο κύριος Φερνάντες. Έχετε σχόλια? Όχι. Άρα... Να ψηφίσουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν έχω μαζί μου κάρτα. Θα προσθέσουμε την ψήφο μου. Η κυρία ε, ούτε και εκείνη. προσωμείωση. Δύο ψήφοι επιπλέον λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμή, τεστ. Δεν έχουμε απαρτία. Καλά, καλά. Άρχεται η ψηφοφορία για επαλήθευση. Άρχεται. Ηλεκτρονική λοιπόν ψηφοφορία, ε, πραγματική αυτή τη φορά, άρχεται. ψήφισαν άπαντες 12 προς 1 από 13 σύνολο, δηλαδή 15. Δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν άλλα θέματα, άρα να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας προβλέπεται στις 10 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο Α, στι 16 και 45. Στις 4 μάλλον. Μπουτ και Έκον. Μετά στο Στρασβούργο. Θα βρούμε το ωράριο αργότερα και 13 Δεκεμβρίου κοινή πάλι με την ΕΚΟΝ στο Στρασβούργο. Και τώρα να δώσω την Προεδρία στον κύριο Σαβαρμά. Σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να με την καταστήσετε, διότι το βράδυ πρέπει να είμαι στο Παρίσι. Θα τα πούμε αύριο, συνάδελφοι.